ως Ελνοκ. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τα πρακτικά της ε, χτεσινής ε, συνεδρίασης είναι στην διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά. Εάν όχι, τότε εγκρίνονται. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε τα κατεπήγοντα που αφορούν τις περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Πρώτο ζήτημα είναι η κατάσταση στο Τζιμπουτί. Τον λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ως ένας από τους λίγους βουλευτές που έχει εμπιστευτεί το Τζιμπουτί πρέπει να πω πως έχει πάρα πολλά θετικά. Ε, είναι ένας θαυμάσιος συνδυασμός γαλλικής και σομαλικής κουζίνας και πολιτισμού στην Ερυθρά θάλασσα. Αλλά υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην διακυβέρνηση και η αυταρχική ηγεσία συχνά καταπνίγει τις θεμελιώδεις ελευθερίες ε, ειδικά των πολιτικών αντιπάλων. Ως εισηγητής για το κέρας της Αφρικής ε, θεωρούσα πως θα πρέπει εκεί πέρα να δικοδομηθούν πραγματικά δημοκρατικοί θεσμοί και οι αρχές να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Έτσι έχουμε σοβαρές ανησυχίες για την εκτεταμένη νοθεία των τελευταίων εκλογών, για τη βία εις βάρος των διαδηλωτών και για τη συνεχιζόμενη κράτηση 60 πολιτικών κρατουμένων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία είπαν οι παρατηρητές των εκλογών που θεωρούσαν τις εκλογές διαφανείς και σημείωσαν πως ήταν οι πρώτες εκλογές που είχαν πολλούς υποψηφίους της αντιπολίτευσης που είναι κάτι θετικό. Αυτό οπωσδήποτε είναι θετικό για το μέλλον, αρκεί οι αρχές της χώρας να δεσμευτούν για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και σοβαρές αλλαγές. Το Τζιμπουτί είναι μια μικρή χώρα η οποία μπορεί να ανθίσει και αξίζει την στήριξή μας. Έχει συνεισφέρει ε, σημαντικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας. Υπάρχουν βάσεις ε, της Ιαπωνίας, των ευρωπαϊκών χωρών, η Αταλάντα συχνά ναυλοχεί εκεί πέρα και βεβαίω πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα, αλλά αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από διπλωματική πίεση για να ε, υπάρξει και δημοκρατία και αντιπολίτευση. Και βεβαίως ε, σε σύγκριση με την ε, Σομαλία έχει αποδειχθεί πολύ πιο επιτυχημένη χώρα και ελπίζω Σομαλία, Σομαλιλάνδη και Τζιμπουτή ε, το κέρας ολόκληρο της Αφρικής να είναι μια μέρα ασφαλής, ανεξάρτητες ε, χώρες που θα ευημερούν και ελπίζω να βοηθήσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κίλ Νίλσεν τώρα για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Στο Τζιμπουτί κάθε πολιτική αντίρρηση ή κοινωνική αντίρρηση ε, απαγορεύεται. Και ένα θέμα είναι ταμπού οι βιασμοί των γυναικών αφάρ που γίνονται από το 1990. Ούτε το Υπουργείο για την, προστασία, την πρόθεση των γυναικών, κανένας δεν τολμά να του καταγγείλει στην ΕΙΦΟΡ. Στο Τζιμπουτί ο βιασμός χρησιμοποιείται ω ένα όπλο πολέμου, ώστε να περιοριστεί και να μειωθεί η ταυτότητα των κοινοτήτων. Στις συμφωνίες ειρήνης ε, του 1994 και του 2001, όπου υπήρχαν διάφορες τραπέζια τραπέζι διαπραγματεύσεων, οι βιασμοί, αυτό το έγκλημα πολέμου παραμένουν ε, στο σκοτάδι και εμποδίζουν κάθε δυνατότητα εθνικής συμφιλίωσης. Ε, το ψήφισμα του ΟΗΕ και το δικό μας καλεί τα κράτη να γράψουν τα σεξουαλικά εγκλήματα στο Σύνταγμα τους αλλά και στην ομοθεσία τους. Η ατιμορρησία για τους βιαστές ε, βασιλεύει στο τσιμποτή. Αυτό που λείπει είναι μια πραγματική πολιτική βούληση. Οι γυναίκες παρά την ε, καταπίεση και την τροπή που νιώθουν είχαν το θάρρος ε, να κάνουν να μήνυση. Συχνά όλα αυτά μπαίνουν σε ένα σιρτάρι και δεν δίνεται συνέχεια. Περιμένουν μια υποστήριξη από πλευρά μας για να τις βοηθήσουμε να καταδικαστούν οι εγκληματίε αυτοί. Τίποτα δεν είναι πιο τρομερό για αυτέ τι γυναίκε θύματα παρά η άρνηση δικαιοσύνη. Χωρί δικαιοσύνη, καμιά νοικοδόμηση δεν θα είναι δυνατή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριο Πρέντα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χώρα αυτή είναι σημαντικός σύμμαχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ομελών της ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας ε, στο κέρας της Αφρικής. Η κατάσταση αυτής της χώρας πέρασε από την περνά από την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Είναι αλήθεια πως η κατάσταση του τύπου στη χώρα όπου οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα τη συγκρίνουν με μια μαύρη τρύπα των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ανησυχητική, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε τα όσα έγιναν στο Τζιμπουτί τους τελευταίους τρεις μήνες μετά από τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές της 22ης ε, Φεβρουαρίου. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα βήμα μπροστά στη δημοκρατική πορεία του Τζιμπουτή, με τη συμμετοχή δηλαδή της αντιπολίτευσης για πρώτη φορά στις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές από τότε που ο Ισμαήλ Ομάρ Γκουελέ ανέλαβε καθήκοντα, οδήγησε σε πολύ ανησυχητική ε, κατάσταση, η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων από την αντιπολίτευση οδήγησε σε, βία καταστολή των ε, διαδηλώσεων και σε σύλληψη αλλά και καταδίκη πολλών ε, ηγετών της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, η δημο... Υπήρχαν πολύ σημαντικέ υποψίες νοθεία. Τέλο, η ελευθερία έκφραση είναι πολύ ευάλωτη στη χώρα αυτή και έχει περαιτέρω επιδεινωθεί, ενώ δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι πρόσκειται στην αντιπολίτευση είναι καταδικασμένοι και φυλακισμένοι. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ε, ζητήσει από τις αρχές του Τζιμπουτή να πάψουν να ε, καταπιέζουν την αντιπολίτευση να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατούμενους και να ξεκινήσουν να ο διάλογο με την αντιπολίτευση ώστε να τελειώσει, να λήξει αυτή η κρίση. Αυτή ήταν μάλιστα η υπόσχεση του κυρίου Γκάλα την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με τους ε, περιφερειακές ε, οργανώσεις που δρούν στην περιοχή και η καλή μας σχέση με τον Τζιμπουτί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να προωθηθούν μακροπρόθεσμες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τάκουλα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάσταση του Τζιμπουτή είναι πραγματικά ανησυχητική. Μακάρι να μπορούσαμε να επηρεάσουμε το κέρας της Αφρικής ε, να αλλάξει η κατάσταση αυτή αν θέλουμε να βοηθήσουμε ε, στον εκδημοκρατισμό και στην, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτές είναι αρχές βέβαια που είναι πολύ σημαντικές για όλες τις χώρες μέλη θα πρέπει να βοηθήσουμε άμα δούμε την κατάσταση στο Τζιμπούτι τα και τις εκλογές του Φεβρουαρίου τα πράγματα είναι ενισχυτικά, έγιναν κρατήσεις έκτοτε, δεν, ε, δεν έγιναν σεβαστά ε, τα δικαι... ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, έγιναν μαζικοί βιασμοί και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε να τα αποφύγουμε στο μέλλον, να κάνουμε κάτι τι. Ξέρουμε ότι η κουλτούρα που επικρατεί στην ε, κυριαρχή στο Τζιμπουτί είναι το Ισλάμ ε, και ότι είναι δύσκολο να παρέμβουμε αλλά σίγουρα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι για τη βάση ε, στην εκπαίδευση, στα σχολεία ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε ή έπρεπε να είχαμε κάνει στο παρελθόν από εκεί και πέρα χρειάζεται τεράστια πολιτική πίεση για την ε, αλλαγή νοοτροπίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών αν απλώς περνάμε ψηφίσματα και στέλνουμε χρήματα δεν, δεν κάνουμε τίποτε χρειάζονται προγράμματα κοινωνικά κοινωνίας των πολιτών χρειάζονται προσπάθειες για αλλαγή της νοοτροπίας για να καταλάβουν οι πολίτες εκεί τι σημαίνει δημοκρατία τι σημαίνει ελευθερία ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους τα ανθρώπινα δικαιώματα και η τήρηση του στο Τζιμπουτή είναι αντικείμενο ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι καταστροφική. Για ορισμένα κράτη-μέλη ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Τζιμπουτί είναι, έχει με, μεγάλη σημασία στρατηγική θέση τρεις στρατιωτικές βάσεις εκεί κλπ κλπ όσον αφορά τώρα το ψήφισμα δεν θα ε, έπρεπε να διορθώσουμε το κομμάτι που λέει ότι οι τρεις βάσεις ε, αποφέρουν κέρδη. Για ποιον όμως για το Τζιμπουτί το αμφισβητώ 40% είναι φτωχή αναλφαβητισμός ε, τεράστιος ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών γυναίκες που βιάζονται που ακροτηριάζονται ε, όσον αφορά τα γενικά τους όργανα ε, άθλια κατάσταση η ανεργία είναι επίσης τεράστια ιδιαίτερα για τους νέους, για τις γυναίκες αλλά αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην αντιπολίτευση και είναι ενάντια στην κυβέρνηση του Μπιτζουτή ε, Έγιναν εκλογές βεβαίως. Για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έλαβε μέρος στις εκλογές. Από το επίσημο, από αποτέλεσμα από τα διάφορα εκλογικά κέντρα μετά την καταμέτρηση δεν είναι γνωστό αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι 100% υπέρ του Προέδρου. Λένε ότι η κατάσταση είναι... Ε, οι εκλογέ ήταν διαφανείς. Νέοι μικρής ηλικία ε, δολοφονούνται στη χώρα αυτή. Ο Νταχέρ Αχμετ Φαρά της αντιπολίτευσης μόλις φυλακίστηκε αυτή τη βδομάδα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την σιωπή σε σχέση με τον Τζιμπουτή. να αφήσουμε τους κρατούμενους να μένουν στη φυλακή. Ο κύριος Δεκέιζερ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο καθένας ε, είδε το Τζιμπουτί όπως ήθελε. Αναφέρομαι στην εκπληκτική ε, γαλλική κουζίνα που ανέφερε ο κύριος ε, Τάνοκ. Να σας θυμίσω όμως ότι σύμφωνα με την ΦΑΟ 180.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Τζιμπουτί χρειάζονται επισητιστική βοήθεια που δεν μπορεί να τη προσφέρει η καταπληκτική αυτή ε, ε, κουζίνα του Τζιμπουτί. Το 21η ε, ε, θέση έχει το Τζιμπουτί όσον αφορά την παραβίαση των, της ελευθεροτυπίας από 179 χώρες. Το Τζιμπουτί είναι πολύ σημαντική χώρα για τη σταθερότητα της Ανατολικής Αφρικής και για μας αυτό δεν μπορεί, πρέπει να μας οδηγήσει σε ασυγχώρητες υποχωρήσεις και το Τζιμπουτί σίγουρα δεν είναι η μόνη η χειρότερη χώρα στο κέρας της Αφρικής. Όμως δεν είναι φυσιολογικό μετά από τις εκλογές του Φεβρουαρίου 2013 οπότε και ζητήσαμε επίγον, κατεπήγον για το Τζιμπουτί γιατί είχαμε αμφιβολίες όπως είπε και η κυρία Βερζιά για την κανονικότητα αυτών των εκλογών που ήταν ειρηνικέ και γιατί ήδη αυτό κάτι είναι αλλά ίσως να υπήρξαν προβλήματα. Από το, 2000, από Φεβρουάριο του 2013 λοιπόν προσπαθούμε να περάσουμε ένα κατεπήγον. Ε, από το 2013 η ΜΚΟ και οι διάφοροι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για πάνω από χίλιους πολιτικούς κρατήμονους. Εγώ θέλω να ε, ακούσουμε τον πρόεδρο του Τζιμπουτή και να τον ακούσουμε με όσα είπε. Μίλησε για αντιπολίτευση. Ε, αυτή τη στιγμή καταστέλλεται αυτή η αντιπολίτευση. Να ασκήσουμε μια πραγματική παραγωγή παρακολούθηση της κατάστασης και ας δούμε αν σε τρεις μήνες, έξι μήνες όντως η επιτυχία του Τζιμπουτή από την πλευρά των διεθνών σχέσεων θα είναι όντως καλύτερα σκορ σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ των ομάδων. Πέτερ Στάσνη, πρώτα απ' όλα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τα βήματα προς τη μεταρρύθμιση όπως το ότι μπορεί και η αντιπολίτευση να καταλάβει έντρες στο Κοινοβούλιο. Τα πολιτικά κόμματα και ο λαός του Τζιμπουτή έχουν επιδείξει δέσμευση για το μέλλον της χώρας τους μέσω της συμμετοχή στις εκλογές. Όμως, ανησυχώ για την τρέχουσα κατάσταση του Τζιμπουτή το οποίο παίζει ρόλο κλειδί στην καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας στην περιοχή. Είμαι εναντίον της καταστολής ε, των πολιτικών αντιπάλων και ζητώ την άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων. Καταδικάζω, κύριε Πρόεδρε, την ε, σεξουαλική βία κατά των γυναικών. Η κυβέρνηση πρέπει να προλαμβάνει τέτοιες λυπηρές πράξεις και να τιμωρεί τους δράστες. Το Τζιμπουτί πρέπει να επιδείξει προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα για, να προωθήσει περισσότερο τις σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλιστές, η κυρία Κρετού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ ενισχυτική στο Τζιμπουτί των όσων συμβαίνουν και με την αντιπολίτευση. Μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου υπήρχε μια ευκαιρία εκδημοκρατισμού της χώρας. Ο πρόεδρος εξελέγει με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, αλλά πρέπει νομίζω να ξεκαθαρίσουν ε, οι μομφές ε, περί νοθείας. Νομίζω λοιπόν πως και η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι διαρχές πρέπει να σεβαστούν τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο βασικότερος δωρητής του Τζιμπουτή οφείλει να χρησιμοποιήσει τη σχέση αυτή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας και επίσης την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και τη θρησκευτικών ακροτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς, ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε στην ομάδα μας ε, το Τζιμπουτί, η θέση του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρη και οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα επίσης το ίδιο είπαν. Τους είχαμε δώσει και το βραβείο ζαχάρο πριν από λίγα χρόνια. Ο Αλέξης Ντετοκβίλ είχε πει πως οι επαναστάσεις ξεσπάνε όταν η κατάσταση βελτιώνεται. Ε, κοιτάξτε, η κατάσταση στο Τζιμπουτί βελτιώθηκε. Και οι εκλογές ήταν ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα, να σταματήσει η βία κατά των γυναικών και ει βάρο των διαδηλωτών. Και πρέπει βεβαίω να τα καταδικάσουμε αυτά, αλλά πρέπει να δούμε και τις θετικέ αλλαγέ που έγιναν. Όμως, θεωρώ πως ε, το ψήφισμα αυτό πρέπει να δείχνει στι αρχέ χώρε πω στηρίζουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για τους Ευρωπαίους Ελευθερίες και ο κύριος Πάσκα. Για ένα λεπτό ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οποιαδήποτε μετάβαση από ένα μονοκομματικό σύστημα προς μια πλουραλιστική δημοκρατία έχει προβλήματα. Και αυτό το αποδεικνύει το Τζιμπούτι. Οι διοικητικέ δομές βεβαίως βασίζονται ακόμα σε ένα μονοκομματικό σύστημα και δεν μπορούν ε, να υποταχθούν αμέσως στην θέληση των πολιτών. Το Τζιμπούτι έχει μια στρατηγική θέση στο κέρας της Αφρικής, γι' αυτό πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση έτσι ώστε να διατηρηθούν ε, να διατηρηθεί αυτή η πορεία προς την δημοκρατία. Οι διώξεις ε, της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης πρέπει να σταματήσουν, ε, οι διώξεις των δημοσιογράφων επίσης πρέπει να εγκαθιδρυθεί κράτος δικαίου και να δοκιμάσουμε μια διαμεσολάβηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για να υπάρξει ένα νέο είδος σχέσεων με ανοχή και σεβασμό η χώρα εξαρτάται από τη χρηματοδότηση ΙΠΑ Ευρώπης και Ιαπωνίας. Εάν συντονιστούμε λοιπόν θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Όμπερμαϊερ από τους μη εγγεγραμμένους. Κύριε Πρόεδρε, το να γίνει βεβαίως μια πρώην απικία δημοκρατική χώρα είναι δύσκολο αλλά αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, μαζικές συλλήψεις, ε, καταστολή της αντιπολίτευσης, καταπίεση των γυναικών, δεν είναι σωστά. Η Ευρώπη δίνει εκατομμύρια ευρώ. Ε, βεβαίως αναγνωρίζουμε πως είναι στρατηγικά σημαντική η χώρα το Τζιμπουτί για την καταπολέμηση της πειρατείας και πρέπει να διασφαλιστεί το εμπόριο στον κόλπο του Άντεν. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα εις, βάρος πρέπει να σταματήσουν να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Σάγια ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση στο Τζιμπουτί σε σχέση ε, με οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημοκρατία δεν είναι καλή δεν έχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να δράσει ελεύθερα έχουν γίνει πολλές ε, συλλήψεις, κρατήσεις υπάρχουν γύρω στους 6.000 ε, πολιτικοί κρατούμενοι Βεβαίω το Τζιμπουτί παίρνει μεγάλα ποσά ω αναπτυξιακή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 50 εκατομμύρια ευρώ πρόσφατα δόθηκαν στο Τζιμπουτί. Ελπίζω εμείς ελπίζαμε ότι τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν στον εκδημοκρατισμό και στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μύρσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ψήφισμα είναι πολύ καλό για την κατάσταση του Τζιμπουτί. Συγχαίρω τους συναδέλφους που το συνέταξαν. Κοιτάξτε, ο, από εκεί και πέρα βέβαια, ο πρόεδρος Γκέλεχ είναι δικτάτορας. Υπάρχουν σίγουρα γίνονται συλλήψεις, κρατήσεις αλλά και πάρα πολλά εγκλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να ληφθούν όλα τα μέτρα και οικονομικής φύσεως κυρώσεις για να ανατραπεί η κακή αυτή κατάσταση του Τζιμπουτή. Ο κύριος Λίσεκ τώρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ίσως θα έπρεπε να επενέσουμε τον Τζιμπουτή για τη βοήθεια που μας παρέχει όσον αφορά την πειρατεία στη θάλασσα και για το γεγονός ότι φιλοξενεί αμερικανικά και γαλλικά και ιαπωνικά στρατεύματα στο έδαφος του να το επενέσουμε επίσης και να το συγχαρούμε για τις προσπάθειες που κάνει για εκδημοκρατισμό της χώρας. Βεβαίως ξέρουμε όμως και τις επιθέσεις που έγιναν ενάντια στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δημοσιογράφους κτλ. Αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να καταδικαστούν και δει στεντορία τη φωνή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να περάσει ένα σαφές μήνυμα στη χώρα αυτή ότι εμείς δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους ε, νοοτροπίες περιμένουμε τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ο κύριος Κέλλη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας έκανε μια πολύ καλή περίληψη για την κατάσταση του Τζιμπουτή Βεβαίως, αν ρωτήσουμε τους πολίτες Ευρώπης που βρίσκεται το Τζιμπουτή πιθανότητα δεν ξέρουν καν που βρίσκεται στον πλανήτη. Είναι κρίμα αυτό γιατί η, θέση γεωγραφική του Τζιμπουτή είναι πολύ σημαντική από στρατηγικής απόψεως. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι από, την, ε, τότε που έγινε ανεξάρτητη η χώρα αυτή προόδευσε ε, και έγιναν και ελεύθερες εκλογές το Φεβρουάριο. Ε, συνεχίζουν όμως να υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό θα πρέπει ίσως να πιέσουμε περισσότερο τα πράγματα ιδιαίτερα σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ κύριο Σταραμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό οι αρχέ του Τζιμπουτί να κάνουν επιτέλου τα απαραίτητα ώστε να πάψουν οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εγγυηθούν επιτέλου τι πολιτικέ, ε, κοινωνικέ ε, ελευθερίε και την ελευθερία του τύπου. Από τι εκλογέ του Φεβρουαρίου 2013, οι διαδηλώσει που αμφισβητούν την νομιμότητα αυτών των εκλογών ε, καταστέλλονται. Θα πρέπει να σταματήσει η των εκπροσώπων τη αντιπολίτευσης και να, επίσης, ε, να σταματήσουν οι βιασμοί και οι ε, ακροτηριασμοί των ε, γυναικών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να πάμε στο Τζιμπουτί για να πάρουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Η ελευθεροτυπία δεν υπάρχει και θέλουμε επιτέλους τα αποτελέσματα των εκλογών να δημοσιευθούν με διαφανή τρόπο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Κόρχολα. Το Τζιμπουτί έπαιξε ρόλο κλειδί στην καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας στο, στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής από την ανεξαρτησία του. Ε, Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η χώρα διανύει μια βαθιά πολιτική κρίση. Όλο ένα και περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν και η κατάσταση του στις φυλακές είναι πάρα πολύ κακή και βέβαια δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει ακριβώς στη χώρα. Ο ΙΕ πέρσι ανέφερε πως 180.000 άνθρωποι χρειάζονται επισητιστική και ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης η βία κατά των γυναικών παίρνει διάφορες μορφές, η βιασμή είναι κοινή, ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών Επίσης είναι σεξουαλική βία η οποία έχει μόνιμη επίπτωση στην υγεία των γυναικών και βέβαια πέρα από την συμφωνία του Κοτονού την οποία έχει συνυπογράψει το Τζιμπούτι έχει, την έχει καταπατήσει. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι του Τζιμπουτή είναι όντως σημαντικός εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωσης, γιατί βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Ε, ε, συνεργάζεται επικοδομητικά στην ε, ε, ε, παγκόσμια σκηνή του Τζιμπουτί και γιατί βρίσκεται εκεί στο στον ε, Ινδικό ωκεανό ε, έχουν ε, εκτελεστεί πολλές ε, Υπάρχουν πολλά έργα και πολλές δράσεις στο Τζιμπουτί, πολύ σημαντικές και βεβαίως ε, είχαν γίνει και διαφορετικές πρόοδοι όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό της χώρας πριν από τις εκλογές του Φεβρουαρίου. Ε, θεωρήσαμε ότι απόδειξη του εκδημοκρατισμού ήταν και το γεγονός ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στις εκλογές και η αντιπολίτευση. Οι εκλογές έγιναν μας λένε καλά. Ωστόσο ε, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση ε, στην καταμέτρηση των ψήφων της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και κρατήθηκαν και εκπρόσωποι, συνελήφθησαν και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Αυτό αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν ε, και γι' αυτό ζητούμε από τον Τζιμπουτί να αναλάβει μέτρα και να κάνει και άλλες προσπάθειες για εκδημοκρατισμό της χώρας και για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι του αντιπολίτευση του Τζιμπουτή άρχισαν επιτέλους ένα διάλογο. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν τους, τις, θα προχωρήσει σωστή πορεία και η, θέλ, πιστεύουμε ότι και θα πρέπει ο διάλογος να υπερέχει της ε, οποιασδήποτε αντιπαράθεσης στη χώρα αυτή για να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα του παρελθόντος για να μπορέσει καλύτερα να συνεργαστεί το Τζιμπουτί με την παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να προχωρήσει το Τζιμπουτί αλλά σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, τις δημοκρατικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει το Τζιμπουτί για να μπορέσει να προχωρήσει και να έχει βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε έξι προτάσεις ε, ψηφίσματος. Οπότε σταματάει εδώ πέρα η συζήτηση. Η ψηφοφόρα από το τέλο τη συζήτηση. Επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη είναι.